Και θα ήθελα παρακαλώ να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε μια σειρά ακροάσεων μετά το κοινότημα της συνεδρίασης, οπότε καλύτερα μην καθυστερήσουμε άλλο. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την κοινή συζήτηση των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ, ΕΜΒΙ και ΤΡΟΑ για την ad hoc αντιπροσωπεία που μετέβει στο Μαρακές 10 με 11 Δεκεμβρίου για την ε, υιοθέτηση του Συμφώνου περί μετανάστευσης. Στόχος της σημερινής συζήτηση είναι να ακούσουμε την ενημέρωση για τη διάσκεψη του Μαρακές και ήθελα να καλωσορίσω την Λίντα Μακάμα, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ξέρω ότι συνεχώς ταξιδεύει και ευχαριστώ που βρήκε το χρόνο και ήρθε. Ε, εγώ δεν ήμουν βέβαια στο Μαρακές, εκείνη ήταν. Εκεί υιοθετήθηκε το σύμφωνο της μετανάστευσης και μάλιστα η Επιτροπή αφιέρωσε πολύ χρόνο και ενέργεια στη συζήτηση αυτού του συμφώνου. Θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τώρα το έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το, τα παγκόσμια σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες ε, όπως κάνουμε από τη διακήρυξη Νέας Υόρκης του Σεπτεμβρίου του 2016. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τη Λότε Κνούτσεν και του συναδέλφου τη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και του εκπροσώπους Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών, του Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση και τη ΥΠΑ τη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για του πρόσφυγε. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότητα τη Λότε που ήταν από την αρχή μαζί μα για τη συζήτηση. Και θα ξεκινήσει. Αυτά από μένα. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Λίντα Μακάβαν. Παρακαλώ, Λίντα. Ευχαριστώ, Κλοντ. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο, πήγα σε λάθος αίθουσα. Και ήρθα από την Σενεγάλη, που άφησα εκεί χειμώνα παραστε, μια επιτροπή παρατηρήση εκλογών και ήρθα στο καλοκαίρι των Βρυξελών. Ε, στο Δακάρ δεν είχε τόσο ήλιο στο καιρό όπως εδώ. Χαίρομαι που ε, με την επιστροφή είδα ηλιοφάνεια για την ενημέρωση τη αποστολή ε, στο Μαρακέ. Ήμουν επικεφαλής τη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη του Μαρακέ για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες, που ήταν διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Φαντάζομαι έχετε λάβει όλοι ένα αντίγραφο της έκθεσης με τον κατάλογο των μελών των διαφόρων πολιτικών ομάδων στην κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Εν συντομία, να σα πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακολουθήσαμε ε, τα εγγένεια, την εναρκτήρια διάσκεψη με την αντιπροσωπεία μας και τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε το λόγο εκ μέρου τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δεύτερη διάσκεψη υψηλού επίπεδου, τη δεύτερη σύνοδο υψηλού επίπεδου και συμμετείχαμε επίσης και στην εκδήλωση για την 70η επέτειο της ε, Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε και πολλές παράπλευρες ε, συναντήσεις. Ε, συναντηθήκαμε με τη Μισελ Μπασλέ, την τη πρόσωπο, με το UN Women, με ε, πρέσβεις από το Μαρόκο και άλλες χώρες και χάρηκα ιδιαίτερα που μου επικεφαλής αυτής της υψηλοπέδου προσωπίας ε, στη διάσκεψη για το σύμφωνο, γιατί το σύμφωνο εξετάστηκε ιδιαίτερο και διεξοδικά ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Μάλιστα πολλέ φορές υπήρχε και παραπληροφόρηση και πολλά fake news. Έλεγαν άλλα αντάλλων μερικές φορές. Ε, χαρακτηρίστηκε ως μυστική διάσκεψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπήρχε μεγάλη παραπληροφόρηση και το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλές χώρες μέλη είτε καταψήφισαν είτε απήχαν. Πάντως στην επίσημη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης που έγινε στην Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, 152 χώρες ψήφισαν υπέρ του συμφώνου, 5 ψήφισαν κατά, η Τσεχία, η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Πολωνία και οι Ηνωμένε Πολιτείε ψήφισαν κατά και 12 χώρες απήχαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Λετωνία και η Ρουμανία. Και μάλιστα η Αυστρία τότε ήταν και προεδρεύουσα στο Συμβούλιο. Από τις, περισσότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Σλοβακία δεν δήλωσε τι ψήφισε. Πάντως όπως και στο παρελθόν, ε, ε, σε αντίθεση με το παρελθόν μάλλον, πρώτη φορά τέτοιες εκδηλώσεις των ΗΠΑ συγκέντρωσαν τέτοια προσοχή. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και κρίμα που δεν το κάναμε για να ενημερώσουμε καλύτερα για το τι εστί σύμφωνο. Πάντω η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έκαναν πολύ καλή ενημέρωση και πολλέ φορέ προσπάθησαν να διορθώσουν τι παρα... παραπλανητικέ πληροφορίε που είχαν κυκλοφορήσει και εμένα. Πάντω ε, και δεδομένου του πολιτικού κλίματο, σε τελική ανάλυση δυστυχώ κυκλοφόρησαν και μάλιστα εσκεμμένα κατά τη γνώμη μου πολλές ε, φαλκιδευμένες πληροφορίες ε, ως των πολέμιων αυτής της διαδικασίας. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την πολυμερή πρωτοβουλία του χαλεπού καιρού που διανύουμε για την πολυμέρεια. Τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Τρει μήνε έχουν περάσει από το σύμφωνο, από την έγκρισή του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και προτείναμε στην έκθεσή μα να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ αυτέ τι διαδικασίε που ξεκίνησαν στην Αμένα Έθνη. Καταρχήν να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή των συμφώνων και να παραμείνουν το σημείο αναφορά και για τη μελλοντική νομοθετική μα προσπάθεια και το μελλοντικό νομοθετικό μα έργο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα οργανωτικά σκέλη ε, και του ε, επόμενου φόρουμ για τη μετανάστευση και να δούμε ε, πώς θα λάβουμε μέρος στο Δεκέμβριο του 2019 στο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες που θα γίνει στη Γενέβη. Οπότε φαντάζομαι το νέο κοινοβούλιο θα πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό, για τη συμμετοχή του. Αλλά καλό θα ήταν να κάνουμε ήδη κάποιο σχεδιασμό στις επιτροπές μας. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ σημαντική παρουσία εκεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλοί εκπρόσωποι πολλών χωρών και εταίροι μας από το νότο, από τις νότιες χώρες, ε, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την μεγάλη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Παγκόσμιο Σύμφωνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ε, συμφωνούμε απόλυτα με την ανάλυση σου. Ήταν πολύ καλή αποστολή και είχαμε και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι πολύ αξιέπαινο το έργο σου, το έργο της αποστολής και πολύ εύστοχη και ανάλυση που μας έκανες. Να περάσουμε τώρα στους καλεσμένου μας από τις διάφορες ε, υπηρεσίες και οργανισμούς. Πρώτα Λότε Γνούτσεν που είναι εκτελεστική διευθύντρια της ΑΕΔ. Παρακαλώ Λότε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Λίντα Μακάβαν και την αντιπροσωπεία σα που μετέβη στο Μαρακέ, γιατί την πραγματικά πολύ κατατοπιστική ενημέρωση που μας έκανε και ευχαριστώ για την ε, στεναρή και απερίφραστη υποστήριξη που επιφυλάξετε στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση. Μια δύσκολη στιγμή και αυτή η δημόσια υποστήριξη σας έκανε τη διαφορά. Και ήταν πολύ σημαντική από θεσμική άποψη αυτή η ε, σημαντική ε, υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του Επιτρόπου Αβραμόπουλου και πραγματικά ήταν σημαντική αυτή η σύσσωμη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο τελευταία στιγμή κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, αλλά ήδη από την αρχή τη διαδικασία δείξατε πόσο προσιλωμένοι είστε σε αυτή τη διαδικασία για τη διαχείριση τη μετανάστευση σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Σα ευχαριστούμε λοιπόν θερμά, κύριε Μαγκάβαν, και Ευχαριστώ και την κοινοβουλευτική αντιπροσωπή που μετέβη στο Μαρακέ. Το σύμφωνο τη μετανάστευση εγκρίθηκε στο Μαρακέ και επίσημα ακυρώθηκε και στη Νέα Υόρκη λίγο αργότερα και έχει γίνει πια πραγματικότητα σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Όπω ξέρετε, δεν είναι δεσμευτικό. Πάντω είναι πηγή έμπνευση ε, και μπορούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό με απτές δράσεις και συνεργασία των διαφόρων εταίρων. Είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή επικοινωνιακή στρατηγική και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό το σύμφωνο και αυτό να το προσέξουμε στην επόμενη φάση που θα δώσει και κάποια συνέχεια. Τώρα, τι θα συμβεί στη δεύτερη φάση έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις, οι προετοιμασίε μάλλον και στη Γενέβη και στη Νέα Υόρκη και η ιδέα είναι το, σύμφωνο, το Παγκόσμιο Σύμφωνο να βελτιώσει τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο για τη μετανάστευση και η προστιθέμενη του αξία είναι ότι δημιουργεί ένα ελαστικό, πολύ ελαστικό πλαίσιο ε, για τη συνεργασία των κρατών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και μπορούν έτσι να σφυριλατήσουν ε, εταιρικέ σχέσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο μεταξύ χωρών, περιφερειών και, να, και χώρες κυρίως προέλευσης για να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που δημιουργεί μετανάστευση. Και στο πλαίσιο αυτό που θα εξετάσουμε ενδελεχώς και στο μέλλον, ήδη πολλά συμβαίνουν και στη, στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί πολλές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που έχουν ληφθεί εδώ και πολλά χρόνια θα είναι ίσως και τμήμα της συνέχειας που θα δώσουμε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο. Τώρα, εμπράκτος, ε, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι στη Γενέβη υπάρχει ένα δίκτυο για τη μετανάστευση που συστήθηκε στα πλαίσια του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, του Παγκόσμιου Συμφώνου. Θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό το δίκτυο και θα έχει στόχο την παροχή συμβουλών σε χώρες που θέλουν ε, πληροφορίες, θέλουν εμπειρογνωμοσύνη και θα πρέπει τα κράτη-μέλη που νιώθουν τέτοια ανάγκη να αναλάβουν πρωτοβουλία για να εξασφαλίσουν αυτή τη συνέχεια για το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη Γενέβη, δημιουργώντα αυτό το κόμβο, αυτό το δίκτυο, το κύκλωμα για τη συγκέντρωση πληροφοριών και εμπειρογνωσία για να βοηθήσουν τι χώρε που θα υποβάλουν σχετικό αίτημα και να τι επικουρήσουν. Και ταυτόχρονα θα έχουμε και ένα μηχανισμό χρηματοδότηση που θεσπίζεται μέσω εθελοντικών συνεισφορών από τα κράτη που ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τις χώρες εταίρους, είτε με τεχνική αρρωγή ή με βοήθεια για ανάπτυξη τεχνικών ικανοτήτων, όπως προβλέπει το σύμφωνο. Υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο σε αυτό το δίκτυο που θα βρεθεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στη Γενέβη, θα υπάρχει και μια γενική πλατφόρμα γνώσης που θα συγκεντρώνει πληροφορίες, ε, στοιχεία και δεδομένα για τη μετανάστευση. Όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται, γιατί ε, ανέκεψη ανάγκη συλλογή πληροφοριών που θα είναι ακριβείς, πραγματικές ε, και θα, αποτελεί, θα αποτελούν σημαντικό τμήμα αυτού του κόμβου, αυτού του δικτύου της Γενέβης. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που βρίσκεται ακόμη στα Σπάργανα να αναπτυχθεί περαιτέρω υπό το συντονισμό, όπως σας είπα, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Και στη Νέα Υόρκη θα δοθεί συνέχεια. μάλιστα, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θα έρθει στην Επιτροπή ΑΦΕΤ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Νέα Υόρκη θα δοθεί μια συνέχεια με έμπρακτο τρόπο και θα πρέπει να θεωρηθεί μια διαδικασία εν το γίγνεσθε. Δεν είναι κάτι στατικό που τελείωσε. Θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια, μια δυναμική διαδικασία. Θα έχουμε και το Διεθνές Φόρουμ για τη Μετανάστευση που θα είναι εδώ συνέχειες. Εκεί θα είναι ένα φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων, για ανάλυση βέλτιστων πρακτικών, και θα είναι μια επίσης πολυμερής ε, προσέγγιση με τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερομένων. Θα γίνει γύρω στον Ιούνιο με Ιούλιο. Η ιδέα είναι το φόρουμ που θα συνέρχεται κάθε τέσσερα χρόνια για να εξασφαλίζει μια συνέχεια, μια παρακολούθηση, ε, να έχει επαφές με τον ιδιωτικό κλάδο, με τους ενδιαφερόμενους, με κυβερνητικές οργανώσεις, διάφορες περιφερειακούς φορείς, με, το παγκόσμιο, με την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη μετανάστευση και με Εθνικά Κοινοβούλια, προκειμένου να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που θα τις ε, αξιοποιήσει για τις ε, αξιολογήσεις που θα κάνει κάθε τετραετία. Αυτά είναι τα βασικά σημεία πρόοδου. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια διαδικασία που εκπορεύεται από τα κράτη, από τα κράτη. Ε, είναι συνεχής, ε, ελαστική και δεν αποκλεί κανέναν, ώστε και οι χώρες ανάλογα με το βαθμό ενδιαφέροντος και προσήλωσή τους μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο ζήτημα. Πάντως έχουμε αναγνωρίσει την ανάγκη για μια συλλογική ε, δράση προκειμένου να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα όλα αυτά τα θέματα. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση από πλευρά τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Και τώρα έχουμε το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση για να μας παρουσιάσει την κατάσταση πως έχει. Ο κύριος Χέντριξεν, ευχαριστώ. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι ένα πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης για να συνεργαστούν τα κράτη καλύτερα, για να υποφεληθούμε όλοι από τα ωφέλη της μετανάστευσης και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Τα κράτη, λέει το σύμφωνο, θα παίζουν τον ηγετικό ρόλο. Κάθε κράτος θα πρέπει να κανονίσει τις προτεραιότητές, της, προτεραιότητές του, να δει σε ποιους στόχους θέλει να εστιάσει και τι βήματα να πάρει για να εξοπλίσει το σύμφωνο. Επίσης, αναφέρεται η εφαρμογή, οι δράσεις για κάθε στόχο. Συγκεκριμένε προτάσεις για το τι βήματα μπορούν να γίνουν για την εφαρμογή του συμφώνου. Είναι περίπλοκο το θέμα τη μετανάστευση. και γι' αυτό το σύμφωνο λέει ότι πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί οικοδόμησης μηχανικού, ούτω ώστε να υπάρξουν διμερεί, περιφερειακές και διεθνεί συνεργασίες για το θέμα αυτό. Στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών θα έχει τρία συστατικά ο πόλος σύνδεσης, ούτως ώστε να ανταλλάσσονται πληροφορίες και επίσης ε, μία πλατφόρμα ενημέρωσης. Και επίσης ένα ταμείο για startup, για να συνδυάσουμε τους πόρους για την αρχική χρηματοδότηση προγραμμάτων για να εφαρμοστεί από τα κράτη το σύμφωνο. Μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ε, αρχή σε αυτού του ταμείου. Αναμένεται ότι φέτο, τα κράτη-μέλη θα κάνουν μία έρευνα των βασικών στοιχείων της πολιτικής τους για να κανονίσουν ε, πώς θα καταρτήσουν τα εθνικά πρόγραμμα δράσης. Θα παίξουν επίσης ε, ηγετικό ρόλο και για την αναθεώρηση και συνέχιση που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του συμφώνου. Θα υπάρχει και ένα φόρουμ για την ε, μετανάστευση, για τη διεθνή μετανάστευση. Θα υπάρχει λοιπόν μια διακυβερνητική πλατφόρμα για τα κράτη-μέλη και άλλους φορείς για να συζητήσουν την εφαρμογή. Θα συναντάτε κάθε τέσσερα χρόνια από το 2022. Γίνονται διαβουλεύσεις τώρα για τις διαδικασίες ε, και τα στοιχεία του τρόπου λειτουργίας αυτού του φόρουμ πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούλιο ελπίζω. Από το 2020 θα έχουμε διαδικασίες σε περιφερειακό, υποπεριφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Συναντήσεις αυτές θα γίνονται κάθε δύο χρόνια. Το σύστημα των ΗΕ Εθνών θα στηρίξει τη διαδικασία εφαρμογής, συνέχισης και μεταρρύθμισης του Συμφώνου Μετανάστευσης. Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Εθνών δημιούργησε ένα δίκτυο για την ε, μετανάστευση. Με στόχο, μεταξύ άλλων, να υπάρχουν ε, συντονιστικές ενέργειες, στήριξη στα κράτη και τα κράτη-μέλη να έχουν στήριξη από τα Ηνωμένα Έθνη σε κάθε επίπεδο, όπου θα υπήρχε προστιθέμενη αξία. Επίσης θα υπάρχουν συνδέσεις με τις δομές των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα επίπεδα. Το δίκτυο αυτό θα απαρτίζεται από οργανώσεις του νεφελώματος των Ηνωμένων Εθνών. Και ο οργανισμός για τη μετανάστευση εργάζεται προ αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρξουν και αποσπάσει από όλου του οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Θέλουμε να στηρίξουμε και τα κράτη και τις κοινωνίες για να υπάρξει συνεργασία που να καλύπτει όλες τις πλευρές του συμφώνου. Η εργασία μας όμως δεν περιορίζεται στους στόχου του συμφώνου. Θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη γενικά όταν το ζητούν. Θα είμαστε ως οργανισμός για τη μετανάστευση σε στενή επαφή με όλα τα κράτη είτε έχουν υιοθετήσει το σύμφωνο ή όχι. Τα κοινοβούλια παίζουν ουσιώδη ρόλο, ούτως ώστε να βασίζεται η πολιτική μας σε στοιχεία και στις διεθνείς προδιαγραφές. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις ανησυχίες των κοινωνιών σε διάφορα κράτη-μέλη, που βασίζονται σε διάφορα προβλήματα ή και σε φόβους. Παράλληλα με αυτό το σύμφωνο έχουμε και το σύμφωνο για τους ε, πρόσφυγες. Ο συνάδελφός μου από τον Οργανισμό για τους Πρόσφυγες θα πάρει το λόγο αμέσως μετά. Αυτές οι δύο δικασίες είναι παράλληλες και αλληλοβοηθούνται. Θα πρέπει να συντονίσουμε τις προσπάθειες για να ενισχύσουμε τα εθνικά συστήματα, για να αντιμετωπίσουμε τα ε, προβλήματα των μετακινούμενων ατόμων, τόσο ώστε να αξιοποιήσουμε καλύτερα και τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη είτε μέσω του δικτύου μετανάστευσης, είτε μέσω του Οργανισμού Στήριξης του Ασύλου και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η είπατε αρμοστία για τους πρόσφυγες, η Σοφή Μαγκίνε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να σε ενημερώσουμε. Για να σας πούμε τι έχει γίνει για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες. Αναλάβουμε μια πρωτοβουλία στις 7 Φεβρουαρίου, όπου δύο μεγάλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις εδώ στις Βρυξέλλες οργάνωσαν ε, μια εκδήλωση όπου συμμετείχαμε και εμείς και πολλοί άλλοι φορείς και η κυρία Σαρτζεντίνη από το Κοινοβούλιο για να ενημερώσουμε και να συνεργαστούμε με τις μη κάπα είναι συνέχεια λοιπόν αυτή τη προσπάθεια που ήδη κάναμε. Όλοι γνωρίζετε ότι υπάρχουν αυτά τα δύο σύμφωνα. Εγώ τώρα αναφέρομαι στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες που επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι μη δεσμευτικό λειτουργικό μέσο για να συνεργάζονται τα κράτη και προέκυψε μετά από δύο έτη διαβουλεύσεων με πολλούς φορείς και τους ίδιους τους πρόσφυγες, στην κοινωνία των πολιτών και εμά βεβαίω. Θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τι χώρε όπου ζουν οι περισσότεροι πρόσφυγε, διευκολύνοντα περισσότερε επενδύσει και από τι κυβερνήσει και από τον ιδιωτικό τομέα για να ενισχυθούν οι υποδομέ και οι υπηρεσίε που παρέχονται και να είναι λοιπόν προ το όφελο και των ε, προσφύγων και των κοινοτήτων που του ε, υποδέχονται. Ε, επιδιώκουμε να εκπαιδευτούν κατάλληλα, να καταδεχθούν κατάλληλα, ούτω ώστε να βοηθήσουν όσο ζουν σε εξορία και να προωθηθεί επίσης η προστασία του περιβάλλοντος και εναλλακτικέ ενέργειες. Και προβλέπει μέσω επανένωσης οικογενειών, μέσω ανθρωπιστικών θεωρήσεων και ε, μέσω και άλλων μεθόδων να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς, αν και βέβαια η καλύτερη λύση είναι η επιστροφή στις χώρες τους για τους περισσότερους πρόσφυγες, σε συνθήκες αξιοπρέπειας θα δημιουργήσουμε σύστημα συνέχιση. Θα έχουμε ένα παγκόσμιο φόρουμ που θα συναντάται κάθε τέσσερα χρόνια, όπου οι κυβερνήσει και άλλοι θα δεσμεύονται για περαιτέρω μέτρα και θα κάνουν απολογισμό για χρηματοδότηση και άλλε ε, βέλτιστες πρακτικέ και για μετεκατάσταση. Το πρώτο φόρουμ θα γίνει στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στη Γενέβη. Η προπαρασκευή είναι ήδη καθοδόν. και θα φιλοξενηθεί από τον ύπατο εκπρόσωπο για τους πρόσφυγες και τον Γενικό Γραμματέα και την Ελβετία. Ο Γενικός Γραμματέας θα μιλήσει στην ανακτήρια ε, εκδήλωση αυτού του φόρουμ. Ποιες είναι οι προπαρασκευαστικές ε, συναντήσεις εν ώψη αυτού του φόρουμ, αν το ξέρετε. Θα έχει τρία στοιχεία. Συναντήσεις υπουργικού επίπεδου, όπου τα κράτη και άλλοι φορείς θα δεσμεύονται και θα ανακοινώνουν τι θα κάνουν για την εφαρμογή του συμφώνου. Όπως είπε και η Λότε, η διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων δεν αφορά μόνο τις κυβερνήσεις, αφορά και τα κοινοβούλια και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλους. Κατόπιν έχουμε μια πλατφόρμα, πλατφόρμα για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και για να βελτιωθεί η ανταλλαγή. Και επίσης θα είναι και μια δυνατότητα αυτό το φόρουμ για απολογισμό της πρόοδου που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των στόχων ένα χρόνο μετά την επικύρωση από τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να υπάρξουν ε, αναλήψει υποχρεώσεων και σε το περιφερειακό επίπεδο. Θα έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που θα επιτρέπει σε ορισμένου να παίξουν ηγετικό ρόλο για αυτό το πρώτο φόρουμ. Και πριν γίνει η πρώτη προπαρασκευαστική θα γίνουν και άλλε ενέργειε. Από ό,τι κατάλαβα, οι προσκλήσει για τι προπαρασκευαστικέ συναντήσει θα βγουν σήμερα. Με ένα οδικό χάρτη για τι συναντήσει που θα έχουμε στην πορεία και τον Απρίλιο θα υπάρξει και ένα έγγραφο με περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων. Στην προετοιμασία λοιπόν για αυτό το Παγκόσμιο Φόρουμ θα έχουμε τρεις προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τα κράτη-μέλη και άλλους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Πρώτη 29 Μαρτίου, δεύτερη 25 Ιουνίου και η τρίτη στις 14 Νοεμβρίου και οι μερίσει διατάξει και άλλα έγγραφα για τι συνεδριάσει αυτέ θα αποσταλούν εγκαίρω. Η πρώτη προπαρασκευαστική τώρα, 29 Μαρτίου, θα ασχοληθεί με τη διαδικασία ανάληψη υποχρεώσεων και δείκτε για το πώ θα σημειώσουμε την πρόοδο, θα μετρήσουμε μάλλον την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων. Ο οργανισμό μα θα ενημερώσει προφορικά για τι προετοιμασίε για το φόρουμ σε μια συνεδρίαση της ε, Μονίμου Επιτροπής το 2019. Θα σε ενημερώσουμε λοιπόν για όλα αυτά και θα στείλουμε πληροφορίες και στην αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Γενέβη και στο Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο για αυτό το φόρουμ. Θα καταρτήσουμε μία τριετή στρατηγική για τις ε, επανεγκαταστάσεις. Θέλουμε να υπάρξει αυτή η στρατηγική για το 2019-2021. Έχει βοηθήσει πολύ το Κοινοβούλιο για να προωθηθεί περισσότερο θα έχουμε και ένα παγκόσμιο πανεπιστημιακό δίκτυο για να στηρίξουμε το σύμφωνο και μία ομάδα στήριξης για το άσυλο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμεθα με το Κοινοβούλιο, το οποίο και ευχαριστούμε και όλους τους θεσμούς της Ένωσης για τη στήριξη για τα σύμφωνα. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το έργο της ΥΠΑ της και για τις πληροφορίες που μας δώσατε σχετικά με το που βαδίζουμε. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην ε, αποστολή και κάποιοι άλλοι που θέλουν παρόλα αυτά να πάρουν το λόγο, ακόμη και αν δεν πήγαν. να δω λίγο. Έχουμε στις 3.30 τις ακροάσεις μας, οπότε αν μπορείτε δύο λεπτά ο καθένας, Γιούντιτ και Ενρίκε και μετά η Σεσίλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Μακάβαν που ηγήθηκε αυτή τη αντιπροσωπεία. Θέλω να συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν εκεί και είχαμε, που είχαμε την ευκαιρία μετά τη δυσφήμιση, αν θέλετε, αυτού του Παγκοσμίου Συμφώνου. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήμασταν εκεί και εκτιμώ πολύ το ότι εκπρόσωποι του ΟΗΕ μας αφιέρωσαν χρόνο. Κυρία Γκραπίνη, καθίστε σας παρακαλώ γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Μπάς περιπτώσει έλεγα ότι είναι σαφές ότι και ο ΙΕ εκτίμησε το γεγονός ότι ήμασταν εκεί γιατί καταφέραμε και κάναμε και διμερείς επαφές με όλους τους αξιωματούχους. Το πρόβλημα είναι τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Μια διχασμένη Ευρώπη πώς ακριβώς θα υποστηρίξει την πρόθεση αυτού του συμφώνου του Μαρακές. Πώς θα σταθούμε απέναντι στις αφρικανικές χώρες οι οποίες μας λένε ότι έχετε χάσει την αξιοπιστία σας ως εταίροι γιατί δεν μπορείτε ούτε καν με μια ενωμένη φωνή να προσυπογράψετε τις αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτό το σύμφωνο. Όταν μάλιστα το σύμφωνο αυτό μιλά και για επιστροφές πολιτών είναι μια, ένα πολύ ενδιαφέρον σύνολο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Οπότε νομίζω ότι το δύσκολο είναι πώς θα καταφέρουμε να καταστήσουμε λειτουργικό τώρα το σύμφωνο τη στιγμή που η ευρωπαϊκή πλευρά δεν παρέχει την αναγκαία υποστήριξη. Ας μου το εξηγήσει κάποιος. Εγώ έχω προσπαθήσει... Ε, όταν θέλουμε να, αν θέλουμε να πούμε στη Μιανμάρ πώς θα χειριστεί και πώς θα αντιμετωπίσει τους Ροχίνγκα, το σύμφωνο είναι ένα πολύ ε, χρήσιμο εργαλείο. Αλλά ε, είμαστε σε μια θέση μάλλον δύσκολη. Κάπως γελιοποιηθήκαμε. Μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε καταψήφισαν. Όλε οι υπόλοιπε αρνητικέ ψήφοι και αποχέ προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ενρίκε. Ευχαριστώ και καταρχήν ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνατε και για το έργο και την προσπάθεια και της ΑΕΔ και των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν τεράστιες προσπάθειες για να προωθήσουν αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες ή τα δύο σύμφωνα, το ένα για τη μετανάστευση και το άλλο για τους πρόσφυγες. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω ε, την ομιλία της κυρίας Σερχεντίνη. Τι εννοώ. Το, στο τελευταίο στάδιο της ολοκλήρωσης ε, της διάσκεψης του Μερακές ήταν πολύ αρνητικά τα αποτελέσματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καταθλιπτικά, θα έλεγα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν υπέρ των δύο παγκοσμίων συμφώνων και θέλαμε να διατρανώσουμε τη φωνή μας, γιατί ε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η μετανάστευση είναι παγκόσμια και στρατηγική πρόκληση όχι μόνο του παρόντος αλλά και του μέλλοντος και θα στιγματίσει την εξέλιξη του κόσμου και όχι μόνο των χωρών που είναι χώρες προέλευσης ε, των μεταναστών και των προσφύγων. Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι φαινόμενα όλων των υπήρων και μάλιστα ε, ακόμη και εκεί που δεν είναι τόσο έντονη ε, υπάρχει παρόλα αυτά. Παρόλο που μπορεί να μην είναι έντονο, τόσο έντονο όσο σε εμά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι όσοι διαπίστωσαν την αποστασιοποίηση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις μιμήθηκαν απλώς ή άλλες που από ξενοφοβικές, ε, ρατσιστικές, ε, αντιμεταναστευτικές, εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις συμπαρατάχθηκαν με τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες που κράτησαν στάση αποχής που θέλαν να ανοίξουν τα σχήρα τους. Απλώς έδειξε ότι οι αλλες χωρες που κρατησαν σταση αποχης που ήθελαν να ανοιξουν τα σχηρα τους απλως εδειξε οτι η ε, έδειξαν απλώς την έλλειψη αλληλεγγύης ε, με αυτά τα τεχνάσματα που έκαναν. Ε, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το δικό μας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει πια την ευκαιρία να παρακολουθήσει κατά πόσο θα εφαρμοστούν και στην πράξη τα δύο παγκόσμια σύμφωνα, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Αφήνω όμως μια παρακαταθήκη στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε, θα, θα το ευχόμαστε να γίνει μια κινητήριος δύναμη πιέζοντας τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν. Παρόλο που τα παγκόσμια σύμφωνα, επαναλαμβάνω, δεν είναι δεσμευτικά. Γιατί η μετανάστευση, η προσφυγιά είναι φαινόμενα που θα μας συνοδεύουν για μερικές γενιές ακόμη κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ, Ενρίκε, η Σεσίλ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Θέλω να σημειώσω τη σημασία της παρουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μαρακές. Εγώ πάντοτε υποστήριζα την πρωτοβουλία αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ε, το Κοινοβούλιο επιμένει να εμφανίζεται προσωλωμένο στους στόχους του συμφώνου. Θέλω να ευχαριστήσω και να συμφωνήσω και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο πριν από εμένα. Από τη μία πλευρά έχουμε μια κρίση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Πρόκειται για μια πραγματική πολιτική κρίση. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να ε, τονίσουμε και το ρόλο της Κομισιόν, ο οποίος δεν είναι εύκολος. Αν όμως θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσει το ρόλο της στο παγκόσμιο στερέωμα, τότε η Κομισιόν πρέπει να επιτελέσει τον πολιτικό της ρόλο, ιδίως όταν υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν μπορούν ούτε καν να καθίσουν και να συζητήσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή για να δείξουμε ότι η Ευρώπη με όλα τα θεσμικά της όργανα παρακολουθεί και στηρίζει τη διαδικασία αυτή. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει πραγματικά να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει το ρόλο της ως διαμεσολαβητή. Όμως και ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν είναι ίσονο σημασίας. Πρέπει να ε, ενημερωνόμαστε τακτικά. Έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλες προσπάθειες στο θέμα της μετανάστευσης και για την ενίσχυση αυτού του παγκόσμιου συμφώνου για τη μετανάστευση, αλλά μας έχει απασχολήσει ευρύτατα και γενικώ το θέμα των προσφύγων, με μια σειρά από εκθέσεις και νομικές ε, προτάσεις που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε στον κόσμο ότι παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ε, γιατί μας ενδιαφέρουν. Όσον αφορά το σύμφωνο για τους πρόσφυγες, νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε το Δουβλίνο. Προφανώ αυτό είναι εσωτερικό ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να δείξουμε και προ τον έξω κόσμο ότι είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή. Επίση, τα μέτρα με τα οποία θα δοθεί συνέχεια ε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπεριλαμβάνουν το Κοινοβούλιο. Ξέρω, ευχαριστώ Σεσίλ. Η νομοθετική αυτή διαδικασία βεβαίως εντάσσεται οργανικά σε αυτήν την ε, συζήτηση. Συνάδελφοι, πρωτού ξαναδώσω το λόγο στην Λίντα. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Όχι. Εντάξει. Λίντα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που τόνισαν τη σημασία αυτής της διαδικασίας και όπως είπε και ο Ενρίκε, η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει με βραχυπρόθεσμες λύσεις. Για τις ε, αναφορές στα βρετανικά μέσα που ανέφερε η Λότε Κνούτσεν. Για την έκθεση της Αφρικανικής Ένωσης όπου αναφέρθηκε ότι δεν θέλει η Αφρικανική Ένωση πλέον να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ε, ε, μετανάστευσης, ιδίως όσον αφορά αυτές τις πλατφόρμες αποβίβασης. Έγιναν λοιπόν κάποιες αναφορές ε, στα Βρετανικά μέσα το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχει, αν έχει η Λίντα κάποια άποψη γι' αυτό θα με ενδιέφερε πολύ. Μπορώ να σας, να σας τα στείλω κιόλας. Ξέρω ότι έγινε και μια σχετική συζήτηση ε, με τους, ε, στη συνάντηση με τους επικεφαλείς ε, των κυβερνήσεων, οπότε δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μου πεις. Ε, πρόεδρος, δεν ξέρω πώς ακριβώς πρόκειται να το κάνουμε. δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους προσκεκλημένους μας να απαντήσει στα αυτά που ακούστηκαν, αλλά από εσάς εξαρτάται. Δεν θέλω να, να πιέσω. Αν όχι, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση. Νομίζω ότι ε, σκοπός έτσι κι αλλιώς ήταν να γίνει μια ενημέρωση, όχι να γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση. Να ευχαριστήσω την Λότε, τη Λίντα, όλους τους συναδέλφους που ε, επισκέφτηκαν το Μαρακές, όλους εκείνους που προσπάθησαν να πάνε στο Μαρακές, καθώς και όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και που συνέβαλαν με στοιχεία και πληροφορίες στη συζήτηση και θέλω να ευχαριστήσω και τους συντονιστές ε, για τα οργανωτικά μέτρα που έλαβαν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τις, τους φορείς ε, που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες. Είναι ε, μια δύσκολη διαδικασία, περίπλοκη, χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα δύσκολα καθήκοντα. Judith, είπες και εσύ ε, ποια είναι τα προβλήματα. Υπάρχουν ε, και πολιτικού χαρακτήρα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Είναι σημαντικό το ότι έγινε σήμερα αυτή η συζήτηση και αυτή η ενημέρωση. Λίντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, η Λίντα θέλει να μιλήσει στους συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η συνεδρίαση μας θα συνεχιστεί στις 15 και 45 στο, στην αίθουσα 6Q2. Ακριβώς πάνω από εδώ δηλαδή. Α, και τέλος. Ίσως είναι η τελευταία κοινή συνεδρίαση που θα έχουμε σε αυτή τη θητεία. Ε, φαντάζομαι, ε, πολλά γίνονται, Brexit, ε, οι συζητήσεις συνεχίζονται. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω με αυτή την ευκαιρία τους συναδέλφους από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και, τους, ε, και το προσωπικό βεβαίως. Ευχαριστούμε Λίντα και σένα και το επιτελείο σου και πραγματικά ήταν πολύ αγαστή συνεργασία που είχαμε για πολλά θέματα. Θα συγκινηθώ τώρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφοι για τη βοήθειά σας. Στις 3.30 θα αρχίσουν οι ακροάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Οπότε ραντεβού και πάλι στις 3.30.